και τρίτων κρατών με διαδικασία η οποία θα εμπλέκει και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προς το συμφέρον των πολιτών μας σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σόλτς. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχει κλείσει η κοινή συζήτηση για τα θέματα αυτά των χρηματοδοτικών εργαλείων και σήμερα στις 11.30 θα γίνει η ψηφοφορία για τα θέματα αυτά. Ακολουθεί ως επόμενο σημείο της μέσης διάταξης η έκθεση του κυρίου Φλόρενς η ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα. Μιλάει πρώτος ο κύριος Φλόρενς ως εισηγητής. <clears throat> Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα καταρχήν να εκφράσω την ικανοποίησή μου έναντι της Κομισιόν η οποία εξεσφάλισε μια πολύ καλή συνεργασία παρά το γεγονό ότι είναι δύσκολο το θέμα αυτό και θέλω επίσης να ευχαριστήσω και όλους αυτούς οι οποίοι συνεργάστηκαν μαζί μου για το θέμα αυτό. Όταν μιλάμε για ηλεκτρονικά απόβλητα δεν μιλάμε μονάχα για παγκόσμια πρότυπα αυτό είναι το ένα μονάχα τμήμα του προβλήματος. Το άλλο τμήμα του προβλήματος είναι και το πώς θα μπορέσουμε εμείς να εξασφαλίσουμε πρώτες ύλες στην Ευρώπη. Ξέρουμε ότι στο προσεχές μέλλον θα έχουμε προβλήματα με την απόκτηση πρώτων υλών για τη βιομηχανία μας <clears throat> και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε και από την οπτική γωνία αυτή την έκθεση της ανάκτησης πρώτων υλών και εδώ βλέπουμε ότι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Συλλέγουμε και ανακυκλώνουμε με τρόπο πολύ διαφορετικό στην Ευρώπη. Οι καλύτερες είναι οι χώρες της, του Βορρά, 16 κιλά το, το άτομο. Οι χειρότερες χώρες, ένα κιλό το χρόνο μονάχα συλλέγουν για ανακύκλωση. Πρέπει να μπορούμε κάποια στιγμή να κατονομάσουμε και να επονιδίσουμε και αυτούς οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα για να συλλέγουν βασικά υλικά. Και αυτό πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα περιλαμβάνεται στι κατευθυντήρε γραμμέ μα. Μέχρι στιγμή ο καθένα κάνει ό,τι του κατεβαίνει, ο καθένα ορίζει του δικού του στόχου και δεν υπάρχει τρόπο να φέρουμε ενώπιον του δικαστηρίου αυτού οι οποίοι δεν τηρούν του στόχου ανακύκλωση γιατί ακριβώ δεν υπάρχουν κοινοί κανόνε. Αυτό πρέπει να αλλάξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μια εσωτερική αγορά εδώ πέρα. Φαίνεται σαν να το κάναμε μόνο χθε αυτό σε ορισμένου. Η εσωτερική αγορά μα φέρνει πραγματικά μεγάλα πλεονεκτήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία δεν πρέπει να τα απαρνηθούμε. Γι' αυτό το λόγο είναι απαραίτητο αυτοί οι οποίοι έχουν δημιουργήσει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο είναι σαν τη γραβιέρα να καταλάβουν ότι είναι απαραίτητο να έχουμε μια συνεκτικότητα. Και γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από την Κομισιόν να εργαστεί περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν για να γίνει πραγματικότητα μια κοινή αντιμετώπιση. Και η χώρα μου δεν είναι ιδιαίτερα η καλύτερη στα θέματα αυτά, αλλά όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να συμβάλλουν στο να υπάρχει μια κοινή δράση για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους ανακύκλωσης πρέπει και οι στόχοι συλλογή και ανακύκλωση να γίνονται πιο σαφεί και να οριστούν με πιο σαφή τρόπο. Επίση πρέπει να παρεμποδιστούν οι παράνομε εξαγωγέ. Όταν ελέγχθηκαν 450 containers με υλικά ηλεκτρονικά τα οποία πήγαιναν για εξαγωγή, 350 από αυτά τα εμπορευματοκιβώτια είχαν παράνομες εξαγωγές. Είναι <clears throat> προϊόντα που περιλαμβάνουν ε, μεγάλες ποσότητες λευκοχρήσου και χρυσού, ιδίως στα τυπωμένα κυκλώματα των υπολογιστών. Πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε καλύτερα τις οικονομικές επιπτώσεις της έλλειψης πολιτικής μας και να έχουμε ένα πλήρες σύστημα για την επιστροφή αυτών των ε, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξοπλισμών και όχι να πετάγονται χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη το τι γίνονται στη συνέχεια. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι πιο εύκολο να δίνουμε πίσω στους ε, παραγωγούς τα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά απόβλητα και όχι απλώς να τα πετάμε στα σκουπίδια. Και ο στόχος μας είναι επίσης να εμποδίσουμε πλήρως τις παράνομες εξαγωγές αυτών των προϊόντων. Σήμερα όταν παράγεται ένα <clears throat> λαμπτήρα, κυρία Πρόεδρε, πρέπει να το, να το, να το δημοσιοποιήσετε σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υπάρξει η έγκριση αυτού του προϊόντος. Αυτό δεν βοηθάει, πρέπει να γίνει πιο απλή και πιο ελκυστική αυτή η διαδικασία. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Φλόρενς. Για την Κομισιόν τώρα έχει τον λόγο ο Επίτροπος κύριος Ποτότσνικ, παρακαλώ. Καλημέρα, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο και τον κύριο Φλόρεντς και την ομάδα του, τους κοιόδες και την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας. Το ενδιαφέρον που υπάρχει για αυτό το θέμα αντικατοπτρίζει τις τροπολογίες που υιοθετήθηκαν και κατατέθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες. Χαίρομαι που πολλές τροπολογίες υποστηρίζουν πλήρως τις ε, προτάσεις Κομισιόν για την οδηγία ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Δηλαδή να εκμεταλλευτούμε πλήρως ε, τα περιβαλλοντικά ωφέλη της οδηγίας με φιλόδοξους στόχους ανακύκλωσης και ανάκτησης που θα είναι ρεαλιστική για όλα τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, να ενισχύσουμε την εφαρμογή και την επιβολή με το να ορίσουμε λεπτόμερους ε, κανόνες για να καταπολεμηθούν οι παράνομες εξαγωγές και να μειώσουμε το αχρίαστο διοικητικό βάρο για του Ευρωπαίου παραγωγού μέσω τη ενισχυμένη συνεργασία εθνικών αρχών. Με το να ενισχύσουμε αυτή την οδηγία μπορούμε να συνεισφέρουμε στο να γίνουμε μια κοινωνία που θα ανακυκλώνει αποτελεσματικά του πόρου τη. Μιλάμε για τον τομέα και των αποβλήτων που αναπτύσσεται ταχύτερα στην Ευρώπη και έχει πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες στο να μειώσει την εξάρτησή μας από πάρα πολύ σημαντικές πρώτες ύλες. Ε, με βάση λοιπόν τη συμφωνία Κομισιών και Κοινοβουλίου θα ήθελα να φέρω κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Στόχοι συλλογής. Χαίρεται η Κομισιόν για το ότι το Κοινοβούλιο αποδέχεται πλήρως τις φιλοδοξίες μας για τα επίπεδα συλλογής. Είναι φιλόδοξο για να υποφεληθεί το περιβάλλον και η αποτελεσματική χρήση πόρων και είναι εφικτό για κάθε κράτος μέλος, κάτι το οποίο είναι επίσης σημαντικό. Η Κομισιόν προτείνει να οριστεί ο τρόπος με νέο τρόπο, με το να αναφερθεί ρητός ε, ως ποσοστό των παραγόμενων αποβλήτων. Συμφωνούμε αρκεί να οριστεί βεβαίως μια αναλογή μεθοδολογία και εμείς θα φροντίσουμε να συνεισφέρουμε στην κατάρτιση αυτή τη μεθοδολογία όπως προτείνει η Αρμόδια Επιτροπή. Επίσης προτείνεται να καταργηθεί ο σύνδεσμος με τα ROX σε αυτή την οδηγία. Βεβαίω το δεχόμαστε γιατί δεν ήταν αυτό ο σκοπό μα. Τέλο, για τα φωτοβολταϊκά, ένα συγκεκριμένο ζήτημα εντό πεδίου εφαρμογή, όπω ξέρετε, είναι τα φωτοβολταϊκά προτείνουμε να εξαιρεθούν ρητός από το πεδίο εφαρμογή οδηγία και αυτό συμφωνεί με, την, ε, με τις προτάσεις της Επιτροπής. Όμως γνωρίζουμε τον αυξανόμενο αριθμό ανησυχιών που υπάρχει ε, όσον αφορά την ε, διάθεση και την τοξικότητά τους. και μια εθελοντική συμφωνία του κλάδου συμφώνησε στο να τηρήσει κάποιες προδιαγραφές και θα δημοσιευτεί πάρα πολύ σύντομα. Πρέπει οπωσδήποτε να αξιολογήσουμε την ε, περιβαλλοντικές επιπτώσεις της διάθεσης των Ιακών πάνελ πριν αποφασίσουμε για τη συμπερίληψή του στην οδηγία. Καταλήγοντας, η νέα οδηγία όπως ξέρετε είναι στη διαδικασία της ε, αναδιατύπωσης, δηλαδή έχουμε κωδικοποίηση υπάρχουσας νομοθεσίας με κάποια νέα στοιχεία και πιστεύουμε πως στη διαδικασία αναδιατύπωσης θα πρέπει επί της αρχής να σεβόμαστε τους συμφωνημένους κανόνες της διαδικασίας. Μόνο αυτά τα στοιχεία έχουν αξιολογηθεί ως προς τον ακτύπητο αλλά συμφωνούμε με τις προθέσεις και την κατεύθυνση κάποιων τροπολογιών που έχουν κατατεθεί από την Επιτροπή θα ήθελα λοιπόν να ακούσω τώρα την δική σας συζήτηση επί της πρότασης και τις τροπολογίες σας και θα επανέλθω με τις ελικές μου παρατηρήσεις. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να είμαι στους ομιλητές εξ των ομάδων για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Θα μιλήσει ο κύριος Ζέμπερ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Καρλ Χάιτς Φλόρενς για την πραγματιστική του προσέγγιση για το ζήτημα αυτό και συγχρόνως θα ήθελα <clears throat> να απαντήσω και να θέσω και ένα ερώτημα προς τον κύριο Επίτροπο. Είπατε κύριε Επίτροπε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα κράτη-μέλη ώστε να αυξήσουν τις ικανότητές τους για την συλλογή αποφλήτων. Αλλά δεν μπορεί μια χώρα να συλλέγει 16 κιλά κατά κεφαλή και άλλη ένα κιλό. Αυτό, μια διαφοροποιημένη λοιπόν αντιμετώπιση είναι λανθασμένη ερμηνεία της πολυμορφίας. Θα πρέπει να είστε πιο αυστηρός με τα κράτη-μέλη στον τομέα της συλλογής αποβλήτων. Δεν μπορούμε να έχουμε ωραίους κανόνες εδώ, τους οποίους δεν τους εφαρμόσουν καθόλου τα κράτη-μέλη. Είδα την ε, ε συνέντευξη τύπου που δώσατε όπου είπατε ότι η Ιταλία δεν έχει καθόλου ακόμα σχέδια για να εφαρμόσει τη συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρικών αποβλήτων. Αλλά η Κομισιόν ως θεματοφύλακας τη συνθήκη είναι υποχρεωμένη να αναλάβει μέτρα. Εδώ πρόκειται για μια ταχαίως αναδυόμενη αγορά και συνδέεται με το μέλλον της Ευρώπης να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την συλλογή των αποβλήτων. Πρέπει τα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν του κανόνε. Αν εσεί οι ίδιοι είσαστε χαλαροί, δεν προχωρούμε καθόλου στα θέματα αυτά. Είναι σημαντικό να έχετε <clears throat> ε, κανόνες οι οποίοι θα είναι λογικοί και πραγματιστικοί και οι οποίοι θα πείσουν και τους καταναλωτές να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την εφαρμογή αυτών των μέτρων, κυρίως τα κράτη-μέλη, θα πρέπει να αναλάβουν πλήρως τις ευθύνες τους για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ζέμπερ. Για τους σοσιαλιστές έχει το λόγο η κυρία Φαν Μπρέμπτ για μισή λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε κύριε Επίτροπε. Ενώ προετοιμάζουμε την ε, Σύνοδο Κορυφής για την Ενέργεια και δίνουμε ιδιαίτερο βάρος σε αυτό το θέμα, πρέπει αυτές οι ωραίες ιδέες να εφαρμοστούν και στην πράξη και αυτήν η φιλοδοξία του Κοινοβουλίου. Και εκεί πέρα κινούνται οι τροπολογίες μας. Είπατε πως πρόκειται για συλλογή η οποία συνεχώς αυξάνεται και δεν είναι μόνο τα απόβλητα σε κάθε κατηγορία και σε κάθε κρίκο αυτής της διαδικασίας αυξάνονται τα υλικά που πρέπει να συλλεχθούν. Όπως ξέρετε δυστυχώς μόνο ένα στους τρεις ε, ανακυκλώνει και μόνο ένα στα δύο αυτά προϊόντα βρίσκονται εκεί που πραγματικά ανήκουν. Οπότε θα πρέπει να θέσουμε υψηλότερους στόχους, καλύτερους στόχους ανακύκλωσης και θα πρέπει να φροντίσουμε η εξαγωγή των προϊόντων αυτών στον υπόλοιπο κόσμο να σταματήσει επιγόντως. Γιατί θέλουμε τα προϊόντα αυτά να μείνουν εδώ και να φροντίσουμε να παραμείνουν σε εμά οι πρώτες ύλες, αλλά και κυρίως γιατί έχουμε ηθικές και οικολογικές ανησυχίες για το τι γίνεται στις τρι... χώρες του τρίτου κόσμου. Με άλλα λόγια, σαφείς στόχοι και συγκεκριμένοι στόχοι είναι οι στόχοι του Κοινοβουλίου το ανέφεραν οι συνάδελφοι και οι σκιοδησίτες και ο κύριος Φλόρενς, τον οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πολύ καλή συνεργασία και οπωσδήποτε το Κοινοβούλιο θα είναι πάρα πολύ ε, αυστηρό και προειδόπιο εδώ πέρα το Συμβούλιο για να εφαρμοστούν αυτά τα πράγματα στην πράξη. Για τη δική μας ομάδα τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το βάρος που πρέπει να δώσουμε στις παράνομες εξαγωγές. Θα πρέπει επίσης να δώσουμε αγώνα για τις μικρές συσκευές. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κανείς δεν ε, ε, έχει πρόβλημα βεβαίω με τα μεγάλα ψυγεία τα οποία συλλέγονται, αλλά οι μικρές συσκευές ακόμα δεν αντιμετωπίζονται σωστά. Κύριε Επιτροπέ, άκουσα πάρα πολύ καλά αυτά τα οποία είπατε για τα φωτοβολταϊκά πάνελ. Ξέρετε πως η ομάδα μου ε, ήταν κατά της εξαίρεσής τους, αλλά θα, τηρήσω, θα ε, κρατήσω αυτό το οποίο είπατε. Είπατε πως θέμε αξιολόγηση και θα δούμε. Θα το συζητήσουμε αυτό οπωσδήποτε με το Συμβούλιο για την συμπερίληψη των φωτοβολταϊκών Οπότε ζητώ και από τους συναδέλφους να εγκρίνουν το φιλόδοξο κείμενο που έχουμε σήμερα μπροστά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εξ των φιλελευθέρων ο κύριος Παναγιώτοφ. Ε, για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι η Ευρώπη δαπανά άνω των 130 δις ευρώ για να εισαγάγει μέταλλα στρατηγικής σημασίας. Χάρη στη νέα οδηγία μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση αν χειριστούμε το πρόβλημα των αποβλήτων αυτών. Ε, ε, εγκρίναμε την πρόταση με μεγάλη πλειοψηφία στην Επιτροπή μου και θα ήθελα να συγχαρώ τον ε, βασικό εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές, ε, διότι εργάστηκαν με εξαιρετικό τρόπο. Η συμβαστική λύση που θα να ψηφίσουμε σήμερα συνιστά βήμα προόδου προς μια καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην Ευρώπη. Τίθενται νέοι, πιο φιλόδοξοι στόχοι θεσπίζεται ένας νέος μηχανισμός συλλογής των αποβλήτων αυτών. Χάρη, σε αυτά τα δύο νέα στοιχεία ε, θα μπορούμε να εφαρμόσουμε πλέον με αποτελεσματικότητα τη στρατηγική της Ένωσης. Μην ξεχνάτε ότι αυτά τα απόβλητα ενέχουν ε, μέταλλα, ε, το πλατίνα, άλλα μέταλλα τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, να ανακυκλωθούν. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το 2006 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εξε, ε, επέριψαν 350.000 τόνους αποβλήτων δίχως να τα ανακυκλώσουν. Γι' αυτό με τον νέο κανονισμό πιστεύω ότι θα σημειωθεί πρόοδος και η έκθεση συνιστά επίσης πρόοδο και για την προστασία του περιβάλλοντος πέρα από την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση. Ζητώ λοιπόν από τους συναδέλφους να υπερψηφίσουν την πρόταση. Σας ευχαριστούμε για τους πρασίνους. Ο αξιότιμος ε, κύριος Στρεμόπλος για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Με την ε, προσπάθεια αυτή ε, αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα όπου τα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά απόβλητα αυξάνονται ραγδαία και εκτιμάται πως θα φτάσουν τα 12,3 εκατομμύρια τόνους μέχρι το 2020. Η αναθεώρηση της οδηγίας είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να σταματήσει η διαρροή επικίνδυνων ουσιών που οφείλεται στην ελλειπή λειτουργία επίσημων σημείων ε, συλλογής, στη μη ορθολογική διαχείριση και τις παράτυπες μεταφορές. Τα βασικά προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ότι πρώτον ενώ το 65% του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που διατίθεται στην αγορά συλλέγεται χωριστά λιγότερο από το μισό επεξεργάζεται και δηλώνεται. τα υπόλοιπα καταλήγουν στο περιβάλλον ή εξάγονται σε τρίτες χώρες. επίσης το υπάρχον ποσοστό συλλογής των 4 κιλών ανά άτομο το χρόνο ε, απόβλητα ε, οικιακής προέλευσης δεν αντικατοπτρίζει την κατανάλωση σε μεμονωμένα κράτη μέλη και συνεπώς οδηγεί σε πολύ χαμηλούς στόχους για κάποιες χώρες και υπερβολικά φιλόδοξους για άλλες. Τρίτον, υπάρχουν διαφορετικέ διαδικασίε εγγραφή και καταχώρηση των παραγωγών στι διάφορε χώρε. Και τέλο, δεν εφαρμόζονται οι δεσμεύσει. Αυτό που κάναμε ήταν πρώτον, διευρύναμε το πεδίο εφαρμογή σε όλα τα απόβλητα, με ορισμένε εξαιρέσει μόνον. Δεύτερον, ενδυναμώσαμε του στόχου για τη συλλογή το 2016 το 85% των ε, αποβλήτων αυτών θα συλλέγεται. Τρίτον, εξασφαλίσαμε ξεχωριστό στόχο 5% για την επαναχρησιμοποίηση ολόκληρων ε, ηλεκτρονικών ε, και ηλεκτρικών συσκευών. Τα κράτη-μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν επαρκείς πόρους για τη συλλογή των αποβλήτων από τα νοικοκυριά. Πέμπτον, οι λιανοπολιτές θα πρέπει όχι μόνο να παίρνουν πίσω τα απόβλητα αυτά με την αγορά ενός καινούριου αλλά θα πρέπει να συλλέγουν και τα πολύ μικρά σε όγκο. Ε, ακόμη δεν θα απαιτείται ο παραγωγός να κατάγεται από τη χώρα που θέλει να εγγραφεί και τέλος επιδιώκουμε ισχυρή παρακολούθηση των μεταφορών. Πάνω απ' όλα όμως αυτό που χρειάζεται είναι να ενθαρρύνουμε την παραγωγή ανθεκτικών συσκευών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Κυρία Γκέρλινγκ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους τους εισηγητές γιατί είναι το έργο τους στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης. Είναι σαφής η γραμμή τους και επί της αρχής θα τους υποστηρίξουμε αυτό το δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε στην Ευρώπη και χρειαζόμαστε ένα νομοθετικό πλαίσιο, μια οδηγία για να τα καταφέρουμε. Φυσικά θα πρέπει να επεξεργαστούμε περαιτέρω κάποιες λεπτομέρειες. Ε, το κόστος, η ανακύκλωση, η επαναχρησιμοποίηση, η τελική διάθεση δεν είναι πράγματα φτηνά, ούτε και δωρεάν σίγουρα. Ε, ο παράγων πληρώνει. Είναι βασική αυτή η αρχή. Δεν μπορούμε να θεσπίσουμε ένα σύστημα που να αυξάνει το κόστος για τους φορολογουμένους, ε, κυρίως στην εποχή που ζούμε με τις δημοσιονομικές εξυγίανσης. Ε, δευτερευόντως, ε, είναι απαραίτητο να παραμείνει ένα περιθώριο ελιγμών για τα κράτη-μέλη. Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Έχουμε φιλόδοξους στόχους, αλλά μη συγχαίουμε τους στόχους με τη συμμόρφωση. Να μην είμαστε υπερβολικά περιοριστικοί ε, σε σχέση με τις διατάξεις που θα εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη για να επιτύχουν τους στόχους. Θα ήθελα να αναφερθώ επίσης, όπως κυρία Φαν ναι, στις μικρές ε, συσκευές ε, και η οδηγία με τους ε, φιλόδοξους στόχους θα επιτύχει μεγαλύτερα ποσοστά συλλογής αυτών των συσκευών στο μέλλον. Προβλέπουμε υπομονησία στην υλοποίηση της δέσμευσης αυτής. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Εξ ονόματος της ΓΚΟΕ, ο κύριος Βίλς, για δυόμιση λεπτά παρακαλώ. Η κυρία Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ έχουμε όλο και περισσότερα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αρχίζουν να αποτελούν ένα πρόβλημα και για το περιβάλλον και για την ανθρώπινη υγεία. Αναγνωρίζει το θέμα αυτό ο κύριος Φλόρεν στην έκθεσή του και όλες οι πολιτικές ομάδες έχουν τονίσει τη σημασία να υπάρξει μια μεγάλη βελτίωση στα θέματα αυτά στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Χρειάζονται πιο αυστηροί κανόνες για τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα. Πιστεύω αγαπητοί συνάδελφοι ότι θα υποστηρίξετε αυτή την ε, ρύθμιση και αυτό θα είναι η καλύτερη μορφή προστασίας των ανθρώπων στις χώρες στις οποίες εξάγονται αυτά τα προϊόντα. <clears throat> και δεν πρέπει φυσικά να υπάρχει εθελα, εθελοντικός χαρακτήρας στο να παίρνουν πίσω οι παραγωγοί. Πρέπει να μπορούν, πρέπει να είναι υποχρεωτικό αυτό, ιδίως για προϊόντα τα οποία περιέχουν ε, βαρέα μέταλλα όπως το, το κάδμιο. Επίσης, πολλές φορές και τα νανοηλικά μπορούν στη διαδικασία ανακύκλωσης τους να έχουν ένα επικίνδυνο χαρακτήρα για τους ανθρώπους και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις παραμέτρους της ανθρώπινης υγείας. Θέλω να κάνω μια έκκληση προς την Κομισιόν να προχωρήσει σε μια συγκεκριμένη εξέταση για, την, για τα νανοηλικά και να μην χρησιμοποιούνται αυτά, να μην τίθενται σε εμπορία αν δεν έχει αποδειχθεί ότι δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα για την ανθρώπινη υγεία. Εμεί έχουμε καταθέσει και δύο τροπολογίε και θέλουμε την υποστήριξή σα. Είναι οι τροπολογίε 101-102. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την Ευρώπη τη Ελευθερία και τη Δημοκρατία, Ο κύριο Ρώση για ένα λεπτό. Σα ευχαριστώ. Έχουμε ε, πολλά επίμαχα θέματα με το Συμβούλιο και δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε σε πρώτη ανάγνωση παρά μόνο στη δεύτερη ανάγνωση. Μόνο το να υπάρχουν κανόνες οι οποίοι θα υποχρεώνουν τους κατασκευαστές να παίρνουν πίσω τα πεπαλαιωμένα προϊόντα, δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε το ποσοστό ανακύκλωσης το οποίο επιζητούμε, το οποίο πρέπει να φτάσει το 60%. Πώς μπορούμε, εάν δεν το πράξουν αυτά τα κράτη-μέλη, να εξασφαλίσουμε ένα ποσοστό ανακύκλωσης 85% αν ένας καταναλωτής <clears throat> ουσιαστικά τα παλιά αυτά ε, υλικά και τους εξοπλισμούς τα δίνει σε κάποιον άλλο. Πώς μπορεί να έχει την ευθύνη για το τι θα γίνει στη συνέχεια. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο το οποίο θα αντιβαίνει στην αρχή της νομικής ασφάλειας για τους καταναλωτές. Και μπορούμε να οδηγήσουμε σε ρυθμίσεις οι οποίες θα είναι επικίνδυνες και για την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμεί είμαστε κατά του κειμένου τη Κομισιόν. Άλλοι ομιλητέ, ξεκινώντα με τον κύριο Σόνικ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Εμείς Ξέρετε πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε τα ηλεκτρικά και ηλεκτρικά απόβλητα τα οποία αυξάνονται και είναι τα απόβλητα εκείνα τα οποία αυξάνονται με τον ταχύτερο ρυθμό. Από τη μία απειλούν την ανθρώπινη υγεία και βέβαια από την άλλη έχουμε και το ζήτημα των πόρων. Ε, η αναθεώρηση λοιπόν της οδηγίας θα πρέπει να λάβει υπόψη και κάποιους ρεαλιστικούς στόχους για τα νέα κράτη-μέλη όπου οι υπολογιστές, ε, ψυγεία, τηλεοράσεις αντικαθίστανται λιγότερο συχνά από αλλού και η ζωή τους είναι πολύ μεγαλύτερη. Ο ε, συγητής, αντιλαμβάνομαι, θέλει να λύσει το πρόβλημα διατάξεων που δεν ωφελούν πάρα πολύ τα νέα κράτη-μέλη. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθεί υπόψη η διαφορά στις αγορές και στην οτροπία μεταξύ συγκεκριμένων κρατών μελών. Εξακολουθώ να θεωρώ πως ο νέος κανονισμός θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερο βάρος στον πνευματικό έλεγχο της συλλογής και σε πάρα πολλά κράτη-μέλη υπάρχουν παρατυπίες, υπάρχουν ε, ε, χαρτιά τα οποία δεν αντικατοπτρίζουν τίποτα. Γίνεται εμπόριο τιμολογίων, ε, ε, συχνά υπάρχουν παραποιημένα έγγραφα ή λένε πως συνέλεξαν μεγαλύτερες ποσότητες από την πραγματικότητα και δεν υπάρχει επαρκής εποπτεία. Υπάρχει λοιπόν μια ολόκληρη μαύρη οικονομία ανακύκλωσης ε, του υλικού εκτός των σωστών εγκαταστάσεων. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον λόγο τώρα έχει ο κύριος... η κυρία Μακάβαν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Εκεί που ζω εγώ, κύριε Επίτροπε, αν θέλω να ανακυκλώσω τίποτα, πρέπει να τα πάω στο Δήμο, η ίδια Υπάρχουν 4-5 ε, στην πόλη μου. Εάν θέλω να κυκλώσω χαρτί, πλαστικό, γυαλί κτλ. είναι στη γωνία του σπιτιού μου. Εάν είναι για μπαταρίες μπορώ να πάρω τις παλιές μπαταρίες σε οποιονδήποτε σημείο πώλησης. Εάν λοιπόν θέλουμε να αυξηθούν οι στόχοι για ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά αγαθά, Πρέπει να έχουμε τέτοιου είδους συλλογή, να γίνει πιο εύκολο για το κοινό να διαθέσει αυτά τα απόλυτα, ειδικά τα μικρά ε, ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά αγαθά. Όταν ορίστηκε αυτός ο στόχος ήταν τελείως ανεπαρκής και ήταν εύκολο να συλλεγεί κανείς με το να ανακυκλώνει κανείς το ψυγείο βεβαίως. Οπότε χρειαζόμαστε ένα πιο φιλόδοξο στόχο για να κινηθεί η αγορά, για να ξεκινήσουν εταιρείε που θα μπορούν να αφαιρούν τα χρήσιμα στοιχεία από αυτά τα αγαθά. Την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσατε, κύριε Επίτροπε, για τη στρατηγική αποτελεσματική χρήση των πόρων. Αυτή η οδηγία αποτελεί μέρος αναπόσπαστο. Θα πρέπει κάθε κομμάτι ηλεκτρικού εξοπλισμού να συλλέγεται και να ακυκλώνεται, γιατί ε, σήμερα στην Ευρώπη αυτό είναι εξαίρεση, αλλά αύριο πρέπει να γίνει ο κανόνας. Ανέφερε ο Καλχάιντς ε, τους λόγους, έλλειψη ε, πόρων και βεβαίως πρέπει να λειτουργήσει αυτή η οδηγία, αλλιώς δεν τα καταφέρουμε ποτέ. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Κρίς ε, Ντέιβις τώρα για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ε, πρόκειται για να διατύπωση οδηγία, αλλά πολλοί ήμασταν εδώ όταν εκπονείται και η αρχική οδηγία, οπότε καλό είναι να καλύψουμε κάποια κενά επί τη ευκαιρία και να ακολουθήσει η οδηγία τον προσανατολισμό που αξίζει και να δώσουμε και το βάρος που αξίζει σε αυτή την οδηγία. Για την ανακύκλωση θέλουμε να καλύψουμε λοιπόν αυτό το κενό λόγω του οποίου πάνε σε αναπτυσσόμενες χώρες ε, ε, τα, τα απόβλητα ε, στη, στους χήτα δηλαδή των αναπτυσσομένων χωρών. τώρα δεν είναι θέμα ποια τροπολογία θα υποστηρίξουμε. όσοι θέλουν να καλύψουν τα κενά υποβάλλουν τις τροπολογίες και αν θέλουν να προστατεύσουν τους χιτά τους ας έρθουν να μας προτείνουν με ποιο τρόπο. Ε, τώρα, δεν έχουμε κλείσει όλα τα θέματα. Υπάρχουν επιχειρήσει ε, που πουλούν σχετικά φτηνά τι συσκευέ, τα προϊόντα του ε, και δεσμεύουν του πελάτε του με συμβάσει για να αγοράζουν συνεχώ καινούριε συσκευέ και τα ανακυκλώνουν, επανασυλλέγουν τι συσκευέ και μετά σε ένα κλάσμα τη τιμή μεταπολούν αυτέ τι συσκευέ. Οπότε υπάρχει ένας τρόπος για να κινηθούμε, δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε ε, τις ηλεκτρονικές συσκευές για να ξεπεράσουμε και το πρόβλημα των εκτυπωτών με τα, το μελάνι των εκτυπωτών ε, που δεν χρειάζεται. Ε, και ασκείται πίεση από πάρα πολλές επιχειρήσεις ε, γιατί με αυτό το έκρισαν ε, σκόπιμο να καλύψουν τα κενά της οδηγίας και θεωρούνται αναλώσιμες συσκευές όπως εμείς εξάλλου και επίσης ο ορισμός δεν είναι ο ίδιος ορισμός ανάλογα με τη χώρα κάτι θεωρείται ηλεκτρονικός εξοπλισμός ή δεν θεωρείται και οπότε για να καταφέρουμε να επιτύχουμε μεγαλύτερη ανακύκλωση θα πρέπει να αναγωνίσουμε την οδηγία κυρία Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ε, είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση η οδηγία ε, και θέλουμε να επιτύχουμε μια πραγματική αλλαγή σε σχέση με το ποσοστό των αποβλήτων ε, που συλλέγονται για να το πετύχουμε αυτό πρέπει με αρμονισμένο τρόπο να ε, μειώσουμε τη γραφειοκρατία και να ε, ε, έχουμε να ισχύουν οι ίδιες διατάξεις για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης. Τώρα για τους νομικά δεσμευτικούς στόχους για τα ίδια τα κράτη-μέλη θα έλεγα ότι όταν λειτουργεί κάτι αισίως δεν πρέπει να το αλλάζουμε εγώ θα προτιμούσα ένα περιορισμένο πεδίο εφαρμογής ε, για την οδηγία, διότι εάν ε, το διευρύνουμε και τα μη ανακυκλώσιμα απόβλητα ή τα απόβλητα με ε, μακρύ κύκλο ζωής θα καλυφθούν από την οδηγία, αλλά δεν μπορούν να συλλεχθούν με τον ίδιο τρόπο αυτά τα απόβλητα. Λοιπόν, πέρα από το να είμαστε φιλόδοξοι, οφείλουμε πάνω απ' όλα να είμαστε ρεαλιστές και να μην ε, δημιουργήσουμε ένα επιπλέον άθος για τις ε, εντόπιε κοινωνίες. Ε, τώρα ο κύριος Νάταλε για δύο λεπτά. Ωραία. Κινητά, φορτιστές, PlayStation, ψηφιακές μηχανές, θερμόμετρα, ψυγεία, καταψύκτες, τοστιέρες, φούρνοι μικροκυμάτων, ρολόγια, ηλεκτρικές οδοντόκρεμες, DVD, ηλεκτρικές σκούπες, video game, ιατρικές συσκευές, τηλεοράσεις, τηλεκοντρόλ, υπολογιστές, στεγνοτήρες και πλυντήρια. Για να αναφέρω λίγα, γιατί όλες αυτές οι συσκευές οπωσδήποτε θα ακριβίνουν λόγω αυτής της οδηγίας. Και σκεφτείτε πως και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει ακόμη πιο αυστηρή αυτή την νομοθεσία τη στιγμή που ο κόσμος πιέζεται και έχουμε ύφεση. Οπότε σας ενθαρρύνω να αντιληφθείτε λίγο τους σκληρά εργαζόμενου φορολογούμενους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να ανακυκλώσετε αυτό το νόμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Λεκή Πρόεδρο. Ο... Α, έχετε διαδικασία. Χωρίς... Μία, Κύριε Νάταλ, μπορείτε μας... Κύριε μας είπατε ότι η ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων <clears throat> αυξάνει την ε, τιμή του προϊόντος. Αν δεν πρέπει να αναλάβει την, ε, την αντιμετώπιση των προϊόντων αυτών ο παραγωγός, ποιος πρέπει να τα πληρώσει. Αυτή τη στιγμή <clears throat> υπάρχουν οι δημοτικές αρχές και άλλοι φορείς οι οποίοι πληρώνουν αυτό το κόστος το οποίο εσείς λέτε πρέπει να το πληρώνει ο παραγωγός. Μ' αρέσει αυτή η διαμάχη. Αλλά, μα ξέρετε πολύ καλά, όπως ξέρω και εγώ, ποιος θα επομιστεί το κόστος. Θα καταλήξει στον φορολογούμενο. <clears throat> Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια βαθιά ύφεση. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια ύφεση από το 1930. Και μιλάμε για τους σκληρά εργαζόμενους φορολογούμενους. Αυτό πρέπει να γίνει λοιπόν σε εθνικό επίπεδο από πολιτικούς που είναι υπόλογοι. Ενώ η Κομισιόν δεν είναι υπόλογη σε κανένα. Αυτό δεν το δέχομαι. Ο κύριος Φλόρεντς πρέπει να λάβει, θέλει να λάβει το λόγο με μία μπλε κάρτα. Θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ στο συνάδελφο, αλλά δεν τον ξέρω ουσιαστικά γιατί δεν ήταν παρόν στη συζήτηση που κάναμε για τα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά απόβλητα. Αλλά τι θα πείτε στους πολίτες όταν σε πέντε ή έξι χρόνια δείτε ότι οι πρώτες ύλε μας έχουν φύγει και είναι είτε στα σκουπίδια είτε σε άλλες χώρες του κόσμου. Δεύτερο ερώτημα. Διαβάστε κάπως την, την, οδηγία. Δεν λέει πουθενά ότι η ευθύνη είναι του καταναλωτή, είναι πραγματικά του παραγωγού. Θέλουμε εμείς να την κάνουμε πιο αυστηρή την, ε, ε, την οδηγία και θα ήθελα να ακούσω και ποια είναι η απάντησή σας για αυτό το ερώτημα where the cost will end up. πού θα καταλήξει. Το το κόστος. Το πληρώσει, αυτός το πληρώνει πάντα. Δεν ανάγκη να το πει η οδηγία. Ποτέ δεν λέτε, ποτέ δεν λέτε ότι θα ανεβάσετε τους φόρους. Ποτέ δεν λέτε ότι θα πάρετε λεφτά από τον κόσμο. Θα σας πω, με τους δικούς μου υπολογισμούς κοστίζει 50 εκατομμύρια λίρες τη μέρα να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επανέρχομαι σε αυτό το οποίο είπα στον Κρίς. Οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται στο επίπεδο του κράτους μέλους από πολιτικούς που είναι, λογοδοτούν στους εκλογείς. Οι δικοί μου οι εκλογείς δεν μπορούν να απολύσουν επιτρόπους. Αυτό είναι αντιδημοκρατικό και είναι λάθος. Ευχαριστώ. Τον λόγο έχει... Ε, Σουλή για ένα μισή λεπτό. Κυρία Ζουλή, ε, τροπέ το υπενθύμησαν οι συνάδελφοί μου επανειλημμένα ότι την ώρα που η Ευρώπη αναρωτιέται ποια πρέπει να είναι η κοινή τη πολιτική για τον, ενεργειακό, τον ε, ανεφοδιασμό τη ε, σε πρώτε ύλε και σε σπάνια μέταλλα, δεν μπορούμε να παραμελήσουμε την σημασία που έχει η ευφυή επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων μα. Γιατί πρέπει να βελτιώσουμε τη συλλογή του, να αποφύγουμε τη διαρροή, την παράνομη εξαγωγή αυτών των συσκευών. Επίσης να αυξήσουμε το ποσοστό συλλογής ε, και να χτενίσουμε ε, την, ε, το νέο νομοθέτημα γιατί από, ανεξάρτητα από αυτό το νομοθέτημα ούτως ή άλλως τις απολύσεις θα τις υποστεί ο καταναλωτής. Αν θέλουμε να είναι αποτελεσματική η νομοθεσία μας και να το καταφέρουμε, αγαπητέ Καρλ Χάινς, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν εργαλεία που ενδείκνεται να χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή, οι πολιτικέ μα θα πρέπει να εμπλακούν περαιτέρω συγκεκριμένα στην συλλογή και στην ανακύκλωση, αλλά δεν μπορούμε να εκτελονίζουμε τον ίδιο τον ότι επειδή παράγει απόβλητα. Ο πολίτη ε, δεν μπορεί να είναι μόνο θεατής, ε, πρέπει να είναι και ενεργός ε, παράγοντα τη ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα αυτό. Ευχαριστούμε. Τώρα ο κύριος Γκαρντίνη. Κυρία Γκαρντίνη. Συμφωνώ. Συμφωνώ με πολλά από όσα άκουσα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η οδηγία. Θα την υπερψηφίσουμε. Αλλά όμως είμαι πεπισμένη ότι θα πρέπει να εμβαθύνουμε σε ορισμένα σημεία στη δεύτερη ανάγνωση. Εγώ για παράδειγμα προσδοκώ ότι η Κομισιόν θα κάνει μία αξιολόγηση για το ανοιχτό πεδίο εφαρμογής διότι άμα πρέπει να σεβαστούμε περισσότερο το περιβάλλον τότε θα έχουμε κάποιο πρόβλημα στο ανοιχτό πεδίο εφαρμογής διότι ένα κλειστό πεδίο εφαρμογής μας δίνει περισσότερες βεβαιότητες διευκολύνει επίσης την εφαρμογή των διατάξεων Επίσης πρέπει να προσέξουμε τις δαπάνες για τους παραγωγείς, διανομής και μεταπολιτές. Αλλά δεν πρέπει να επιβαρύνουμε όσον αφορά στις διοικητικές επιβαρύνσεις εγώ θεωρώ ότι τα μέσα και τα κριτήρια πρέπει να διαμορφωθούν ανάλογα με το σύστημα της κάθε χώρας. Δεν έχουμε κακές και κακέ καλές και κακές χώρες μόνο, αλλά υπάρχουν και διαφορετικά συστήματα, διαφορετικές καταστάσεις στα κράτη-μέλη που θα πρέπει να αξιολογηθούν ούτως ώστε να μην έχουμε χώρες αυτόματα προνομιούχες και χώρες αυτόματα επιβαρημένες. Χρειαζόμαστε λοιπόν εμβάθυνση. Ο κύριος Πιετικά είναι για ένα λεπτό. Κυρία Πιετικά είναι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, έχουμε μία νέα στρατηγική από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι έγκαιρη η πρόταση αυτή κυρίως ε, για να αντιμετωπιστεί το θέμα των πρώτων υλών ε, τα απόβλητα των ε, μικρών κυρίω ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, των κινητών τηλεφώνων Φερπίν, καταλήγουν στους χιτά τις περισσότερες φορές και κυρίως στους χιτά των τρίτων χωρών όπου αποτεφρώνονται. Ε, ο μηχανισμός αυτός δεν οδεύει προς την ε, σωστή κατεύθυνση, κυρίως ε, μιλώντας για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. το ιδανικό είναι να επαναχρησιμοποιηθούν οι πρώτες ύλες και ελπίζω ότι Ιστερότερα θα είμαστε σε θέση να θεσπίσουμε ένα καλύτερο σύστημα κοινοποίησης καταγραφής σε, σε Μητρώα κατά την εφαρμογή, τη μεταφορά μάλλον της οδηγίας στην εθνική νομοθεσία των ε, κρατών μελών. Ε, προφανέστατα ε, τίθεται και το ζήτημα της διαφοροποιημένης συλλογής που οπωσδήποτε πρέπει να καλύψει η οδηγία. Είναι βέβαια καλό εφαλτήριο η πρόταση οδηγίας. Ελπίζω ότι οι καταναλωτές θα υπομιστούν περισσότερο τις ευθύνες τους στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Γιούζο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι στους στόχους που θέτουμε. Όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε ταυτόχρονα ότι δεν είναι ευκόλως εφαρμοζόμενη η πρόταση του εισηγητή για όλα τα κράτη-μέλη. Παρόλα αυτά βέβαια θα θα υποστηρίξουμε τη θέση του στην πρώτη ανάγνωση η Ισπανική Αντιπροσωπεία. Αυτό το οποίο δεν θα υποστηρίξουμε είναι το εξής. Θέλουμε να υπάρχει μία διάκριση μεταξύ του κόστους της ανακύκλωσης και του κόστους των αποβλήτων. Θα υπερψηφίσουμε την 52, το 1401 και την 1403. Εμείς θεωρούμε ότι οι καταναλωτές πρέπει να ξέρουν τι στοιχίζει αυτή η επεξεργασία και αυτό θα τους επιτρέψει να σέβονται τον νόμο. Επίσης είναι καλό να υπάρχει επαρκής διαφάνεια στην αλυσίδα εμπορευματοποίηση. Ευχαριστώ για το Catch the Μεζάρος. Κυρία Μεζάρος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και σας ζητώ συγγνώμη γιατί άργησα λίγο να σηκωθώ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Φλόρεντς για την εξαιρετική του έκθεση. Μιλούμε για όλο και περισσότερα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Θέλουμε να προωθήσουμε την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, γιατί έτσι θα αλαφρύνουμε και το περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα θα μετριάσουμε και την απώλεια πρώτων υλών, γιατί 85% των αποβλήτων θα συλλέγεται, αλλά μόνο 30% από αυτό το 85% επαναχρησιμοποιείται σωστά. Θα πρέπει να δούμε και τα φορτία των αποβλήτων και να δούμε με την νέα οδηγία αν θα υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Το θέμα της συλλογή αποβλήτων επίσης είναι πολύ σημαντική πρωτοβουλία για να μπορέσουμε να επαναχρησιμοποιήσουμε τις πολύτιμες πρώτες ύλες που διαφορετικά χάνονται. Η ισχύουσα οδηγία δυστυχώς δεν ερμηνεύεται με τον ίδιο τρόπο από όλα τα κράτη-μέλη. Μιλούμε για ταξινόμηση σε διάφορες κατηγορίες, ενώ στην οδηγία μιλούμε για το σύνολο του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογή. Νομίζω ότι ιδιαίτερα στις νέες χώρες μέλη θα πρέπει να έχουμε επιλεκτική συλλογή των αποβλήτων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λίβερ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ζούμε σε μια κοινωνία που παράγει πολλά απόβλητα. Και τα απόβλητα αυτά τα χαρακτηρίζουμε σκουπίδια ουσιαστικά, αλλά μερικές φορές είναι χρυσορυχία όταν μπορούμε να ανακτήσουμε ορισμένες από τις πρώτες ύλες. Δεν μιλούμε για απόβλητα, για σκουπίδια, για απώλεια δηλαδή. Μιλούμε για πραγματικό κέρδος. Θα πρέπει μια και είμαστε πολύ εξαρτημένοι από τις πρώτες ύλες, να μην τις κατασπατάλουμε, να προσπαθούμε να τις επαναχρησιμοποιούμε όσο γίνεται περισσότερο. Εκτός ότι προστατεύουμε και το περιβάλλον. Συζητήσαμε για κάποιες εξαιρέσεις. Είδαμε τι γίνεται με το κάδμιο και τη στρέβλωση ανταγωνισμού υπάρχει μερικές φορές. Επίση θα πρέπει να επενδύσουμε στην καινοτομία και την έρευνα για τη θέση σε εμπορία νέων προϊόντων. Αλλά να εφαρμόσουμε και πιο αυστηρούς ελέγχους στα νάνο απόβλητα. Είναι πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνουν πιο αυστηρούς τους κανόνες για τις εξαγωγές αποβλήτων. Να σταματήσουν οι εξαγωγέ αποβλήτων προ τρίτες χώρε. Ευχαριστώ κύριο Σιρουμπίχη. Ο κύριος Ρούμπιξ. Κύριε Πρόεδρε, είμαι ένα από τα άτομα τα οποία στηρίζουν την ε, ψήφιση αυτής της εκθέσεως και την ε, ξεχωριστή συλλογή ε, αποβλήτων σε αυτή την κατηγορία διότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών παραμένει χωρίς ξεχωριστή διάθεση αποβλήτων και γι' αυτό ανησυχώ διότι σύμφωνα ε, με το σύστημα ε, θα υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ κρατών μελών γι' αυτό και παρακαλώ τα κράτη-μέλη να είναι πολύ προσεκτικά και να ελέγξουν πόσο θα εφαρμοστεί αυτή η οδηγία διότι στην Λετωνία έχουμε περίοδο μέχρι το 2016 για το, και μόνο το 2023 θα έχουμε πετύχει το 65%. Ευχαριστώ. Τον λόγο έχει τώρα ο κύριος Πάσχα. Ε, κυρία ε, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, το θέμα αυτό έχει προκαλέσει πολλή συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, θα, έχουν υποβληθεί και πολλές τροπολογίες. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η συμβιβαστική λύση θα είναι προς όφελος των αποβλήτων. Θεωρώ δε ότι είναι καλό να υπάρχει ε, μία αναμόρφωση του άρθρου 47 κατά τρόπον ώστε το σύστημα συλλογής να ε, στηρίζεται και ε, να μην διαφοροποιούνται οι στόχοι ιδίω στις χώρες όπου δεν υπάρχει η κατάλληλη υποδομή για την διαχωρισμένη ανακύκλωση και διάθεση διάθεση αποβλήτων. Πιστεύω ότι πολλοί από τους εμπόρους αλλά και τους πολίτες δεν εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους και θα πρέπει να βρεθεί ένας εύσχημος τρόπος να λυθεί αυτό το θέμα. Ο Επίτροπος Ποτόκνικ. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλοί από τους ευρωβουλευτές αναφέρθηκαν στην εφαρμογή της οδηγίας που είναι προβληματική. Η εφαρμογή όμως δεν είναι προβληματική μόνο σε αυτό το τομέα. Την αντιμετωπίζουμε σε όλο το περιβαλλοντικό φάσμα των οδηγιών. Γνωρίζω το καθήκον μου όπως απορρέει από τη συνθήκη και θα το ασκήσω πλήρως. Προετοιμάζουμε και μία ανακοίνωση περί εφαρμογής θα κατατεθεί αργότερα μέσα στο έτος που θα πραγματευτεί τα ζητήματα της εφαρμογής με πιο σφαιρικό τρόπο. Το εξετάζουμε με την αρμόδια γενική διεύθυνση γιατί πραγματικά η εφαρμογή είναι ένα από τα ζητήματα που θα πρέπει να μας απασχολήσει στο μέλλον και για άλλες οδηγίες αλλά και για τη συγκεκριμένη. Και μάλιστα η πρόταση αναδιατύπωση σίγουρα διευκολύνει την εφαρμογή. Δεύτερο ζήτημα, οι στόχοι. Νομίζω ότι είναι κεφαλαιόδου σημασία να θεσπίσουμε φιλόδοξους στόχους. Πολύ μιλήσατε για ένα κλάδο αποβλήτων που διωγγώνεται με ταχύτητα τους ρυθμούς γιατί έχουμε όλο και περισσότερα ε, έχουμε όλο και περισσότερες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευέ και άλλο, όλο και περισσότερα απόβλητα. Οπότε θα πρέπει να έχουμε φιλόδοξους στόχους. Για το κόστος. Εμείς στις προτάσεις μας θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το κόστος και ποιον θα επιβαρύνει και θα πρέπει να πλουστεύσουμε αυτές τις διαδικασίες για την επίρρηψη του κόστους. Πάντως θα πρέπει να είμαστε σαφείς. Το πραγματικό κόστος ε, για την κοινωνία και την οικονομία μας ε, θα προκύψει αν δεν είμαστε αρκετά φιλόδοξοι και αν δεν ε, εφαρμόσουμε αυτή την οδηγία. Γιατί μακροπρόθεσμα δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Πριν λίγες μέρες υποβάλαμε μία έκθεση για τα απόβλητα και μάλιστα ε, πραγματοποίησε επίσκεψη σε μία ε, εταιρεία που είναι μία από τις μεγαλύτερες ε, που ασχολούνται με την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και πραγματικά με συγκλώνησαν κάποια στοιχεία που είδα και που διάβασα και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για όλους μας να συνειδητοποιήσουμε ότι τα κινητά που κρατάμε στα χέρια μας καθημερινά περιέχουν πολύτιμα υλικά, πλατίνα, χρυσό. Αυτά τα υλικά είναι πραγματικά πολύ σημαντικά για το μέλλον. Και επειδή μιλούμε και για σπάνι πρώτων υλών, δεν θα πρέπει να αφήνουμε ανεκμετάλλευτα τα απόβλητα, γιατί και αυτά περιλαμβάνουν πρώτες ύλες. Ε, έπιασα 20 κιλά χρυσού που συλλέγησαν από κινητά ε, τηλέφωνα. Ήταν πολύ δύσκολο να σηκώσω αυτό το βάρος των 20 κιλών και ακόμη πιο δύσκολο ήταν να το αφήσω <laughs> κάτω μετά από τα χέρια μου γιατί ήταν χρυσό. Νομίζω ότι θα πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη και το θέμα της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των πόρων. Αυτό το αναφέραμε πολλές φορές, αλλά δεν θα πρέπει να το ξεχνούμε. Θα πρέπει συνέχεια να το έχουμε στο μυαλό μας τον 20ο αιώνα, με βάση στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, ο ανθρώπινος πληθυσμός τετραπλασιάστηκε. Οι 17 φορές δεκαπλασιάστηκαν οι, οι του διοξιδίου, 60 πλασιάστηκαν η βιομηχανική παραγωγή, ενώ πολλαπλασιάστηκαν πολύ περισσότερο από τον πληθυσμό η, κατανάλωση του ύδατος Οπότε δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό. Θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Και χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Γι' αυτό και η πρόταση που έχετε σήμερα χείρας είναι πολύ σημαντική για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Ζητήσατε όλοι καλύτερη διαλογή των αποβλήτων, καλύτερο διαχωρισμό, καλύτερη ενημέρωση. Συμφωνούμε με όλα αυτά και θα ήθελα κατακλείδη να πω ότι μετά την πρώτη ανάγνωση πιστεύω ότι, πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα, σε μια καλή οδηγία και ελπίζω ότι μετά τη δεύτερη ανάγνωση θα διεκπαιρεώσουμε το έργο μας με ένα αποτέλεσμα που θα είναι ακόμη πιο καλύτερο από το σημείο αφετηρίας μας. Ευχαριστώ Επίτροπε. Ο κύριος Φλόρεντς, ο εισηγητής, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ιδίω όσον αναφερθήκατε στα τελευταία σας λόγια στην αποδοτικότητα των πόρων και των πρώτων υλών δεν μπορώ παρά να το υποστηρίξω. Ξέρετε όμως ότι υπάρχει μία εξέλιξη στην Ευρώπη και πρέπει να αποφασίσετε με το Συμβούλιο και στους τελευταίους 7 μήνες δεν έχει κουνήσει ούτε ένα χιλιοστό από την θέση του το Συμβούλιο υπό την ε, ε, ε, Βελγική Προεδρία. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι οι συνάδελφοι οι οποίοι μίλησαν θετικά για αυτή την έκθεση θα πρέπει να επέμβουν και στην κυβέρνησή τους και να πούν ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε όπως ήταν στο παρελθόν. Θα μπορούσα εδώ να αναφέρω διάφορους συναδέλφους οι οποίοι θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν και στους επόμενους μήνες στις συζητήσεις σας θα πρέπει να μείνετε αμετακίνητο στις συζητήσεις με το Συμβούλιο κατά τρόπον ώστε στην πολιτική αποβλήτων ε, να ε, ε, μπορέσει κανείς κάπως να μειώσει αυτή την εθνική νοσταλγία που υπάρχει. Δεν πρέπει να συνεχιστεί διότι εδώ μιλάμε ότι τουλάχιστον το ίμι ε, της εσωτερικής αγοράς υποφέρει 16 προς 11 ε, και φαντάζομαι ότι δεν χρειάζεται να σας δώσω μαθήματα ξέρετε τη δουλειά σας ξέρετε τις ευθύνες σας και θα κάνετε ό,τι μπορείτε για να μας υποστηρίξετε σας ευχαριστώ Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση και θα ψηφίσουμε σήμερα στις 11.30. Διακόπτουμε την Ολομέλεια μέχρι τις 11.30 που ξεκινούν οι ψηφοφορίες.